ότι η μερίσια διάταξη τώρα προβλέπει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου, περίπτωση της Ισπανίας. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στην ε, Σεσίλια Βίλκστρομ, που είναι η συντάκτρια της προφορικής ερώτησης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Η συζήτηση σημερινή και η ερώτηση αυτή προέρχονται από διάφορες αναφορές που πήραμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Αναφορών δηλαδή, τα τελευταία δύο χρόνια και ως μέλος της Επιτροπής αυτής αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά και ειλικρινά θλίβομαι για τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει οι αναφέροντες στην Ισπανία κυρίως, αλλά τέτοια προβλήματα έχουν εντοπιστεί και σε άλλες χώρες μέλη. Η Επιτροπή Αναφορών αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και έτσι ως πρόεδρος της Επιτροπής αυτής θέλω να βοηθήσω τους πολίτες μέσω της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να φροντίσουμε για την καλύτερη εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των ευρωπαϊκών διατάξεων. Διότι πρέπει να βελτιώνουμε την νομοθεσία. Έτσι λοιπόν, με τον ρόλο μας να φέρνουμε τις ε, αναφορές των πολιτών στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνουμε τη συζήτηση αυτή σήμερα, γιατί πρόκειται για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσον αφορά κατάλληλη πληροφόρηση των καταναλωτών σε σχέση με τα ανυπόθηκα δίκαια. Η έγκυρη πληροφόρηση κυρία Πρόεδρε, είναι ζωτική σημασία προκειμένου να μπορέσει κανείς να πάρει σωστές αποφάσεις και είναι ζωτική σημασία όταν μιλάμε για προσωπικές επενδύσεις των ε, πολιτών που έχουν να κάνουν με του ίδιους και με τις οικογένειε τους. Οι αναφορές αυτές μιλούν για πάρα πολλές καταχρηστικές ρήτρες και πρακτικές στον ισπανικό τραπεζικό τομέα που εντοπίστηκαν και από εθνικά αλλά και από ευρωπαϊκά δικαστήρια. Πολλοί πολίτες λοιπόν ήταν θύματα οικονομικών απατών γιατί οι τράπεζες τους πούλησαν ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου χρηματοπιστωτικά προϊόντα χωρίς να τους ενημερώσουν για τους κινδύνους που ελοχεύουν οι επενδύσεις τους. Και δεν έκανε και τις δοκιμές που έπρεπε η τράπεζα για να καταλάβει κατά πόσον οι καταναλωτές είχαν την ικανότητα να αντιληφθούν τον κίνδυνο ή όχι κάτι το οποίο οδήγησε σε φοβερά προσωπικά δράματα και τεράστιες οικονομικές απώλειες. Έχασαν τα σπίτια τους πολλοί πολίτες και τις αποταμιεύσεις μια ζωή ημέρος αυτών. Πολλές τέτοιες τραγωδίες ε, λοιπόν ε, μας τις διηγήθηκαν οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι μπροστά στα μάτια μας στην Επιτροπή να Έτσι λοιπόν με τη σημερινή συζήτηση πρέπει να θέσουμε το ζήτημα σε ένα πλαίσιο. Να φροντίσουμε να υπάρχει σαφήνεια για ένα γενικό πρόβλημα που είναι οι τραπεζικές πρακτικές που τις συναντάμε όχι μόνο στην Ισπανία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρέπει να υπογραμμίσω εδώ ότι η διαφάνεια είναι ε, πολύ βασικό στοιχείο για την προστασία των πολιτών αν θέλουμε να αποφύγουμε καταχρηστικές ε, πρακτικές στον τομέα των ενυπόθηκων δανείων και να προστατεύσουμε τους πολίτες μας. Πάντω, εκ μέρου της Επιτροπής μου, θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια ζητήματα επ' αυτού. Και ελπίζω ότι οι έρευνε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα συμπεράσματά τη θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την κατάσταση όσον αφορά τους αναφέροντες και θα μπορέσουμε να αποφύγουμε στο μέλλον τέτοιου είδου πρακτικέ. Ελπίζω συγχρόνω ότι θα βελτιωθεί και η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αγαπητοί Επίτροπε, λοιπόν, βάσει των αναφορών που έχουμε, πρέπει να απαντηθούν σήμερα τα εξή ερωτήματα. Πρόκειται για παραβίαση της τραπεζικής νομοθεσίας από πλευράς της τράπεζας όταν δεν ενημέρωσαν τους καταναλωτές βάσει της οδηγίας MIFID και βάσει όσο προβλέπει η Ισπανική νομοθεσία. Δεύτερον, η Ισπανία την MIFID 1 την ασωμάτωσε στο εθνικό δίκαιο. Σωστά, οι Ισπανικές αρχές εφάρμοσαν τι σχετικέ διατάξεις. Επίσης ρωτάμε τι μέτρα έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή θα λάβει για να αντιμετωπίσει τις, τις κατακριστικές αυτές πρακτικές που πουλούν χρηματοπιστωτικά προϊόντα σε μικρούς καταναλωτές, όπως για παράδειγμα προνομιούχες μετοχές, που πολλές φορές η διαδικασία αυτή δεν συμμορφωνόταν πλήρως στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Θέλω επίσης να γνωρίζω κατά πόσο η Επιτροπή θα πάρει κάποια μέτρα όσον αφορά το ισπανικό δίκαιο για τα ενυπόθηκα δίκαια και όσον αφορά τις αθέμητες πρακτικές και την μη σωστή συμπεριφορά των τραπεζών που χορηγεί δάνεια στον κόσμο. Θέλω απαντήσεις από την Επίτροπο Γιούροβα και θέλω να ακούσω βέβαια και τους συναδέλφους Και προσωπικά θέλω να σας πω ότι θα πρέπει να δείξουμε κατανόηση στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τόσο πολύ υποφέρει, αλλά θα πρέπει και να διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία στο μέλλον θα είναι ασφαλής και σωστή για όλους στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιούροβα έχει το λόγο, εξ ονόματος της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, καταρχήν θα ήθελα να απαντήσω στις ερωτήσεις 1 και 2. Ναι, πολλοί δανειστές από την Ισπανία βρέθηκαν σε δεινή οικονομική κατάσταση. Υπήρχαν μεγάλα προβλήματα στην αγορά υποθηκών και δυστυχώς ε, οι συμβάσεις αυτές ε, δεν ήταν παρά καταχρηστικές. Και σε αυτή την περίπτωση πολλοί Ισπανοί δικαστές ε, αναφέρθηκαν σε αυτά τα απαράδεκτα ενυπόθηκα δάνεια, τα οποία δεν δέσμευαν τους καταναλωτές. Όπως ξέρετε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ασχολήθηκε με παρόμοια ζητήματα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν υπήρχαν σωστές ρήτρες διασφάλειες προς τους καταναλωτές. Συνεπώς, το ισπανικό δίκαιο τροποποιήθηκε δύο φορές. Μπορεί καταρχήν να προσβάλλει ο καταναλωτής τις καταχρηστικές αυτές ρήτρες των ενυπόθηκων δανείων. Επίσης, το δικαστήριο θα πρέπει να επαληθεύσει αυτές τις συμβάσεις, τα μεταβατικά μέτρα του 93 ε, κάθετος 13 έχουν αμφισβητηθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Επίσης, έχει αποτιμηθεί η ισπανική νομοθεσία και γίνεται ένας διαρθρωμένος διάλογος με τις ισπανικές αρχές. Βασίστηκα στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που θα πρέπει να μεταφερθούν πλήρως στην Ισπανία. Καλωσορίζω τις αλλαγές που έχουν γίνει στην Ισπανία διότι βελτιώνουν την προστασία των καταναλωτών όμως θα πρέπει να προσδιορίσουμε και να δούμε ε, οι ισπανικοί κανόνες σε σχέση με τα ενυπόθηκα δάνεια ε, τηρούν το γράμμα της οδηγίας 93 κάθετος 13 πέρσι τον Ιούνιο αναλύονται τα δεδομένα της Ισπανικής κυβέρνησης από την Κομισιόν και θα δούμε κατά πόσο οι απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές. Σε σχέση τώρα με την πώληση ορισμένων ε, χρηματοπιστωτικών ε, προϊόντων με βάση το υπόμνημα συνεννόησης του Ιουλίου 2012 μεταξύ Κομισιόν και Ισπανίας οδήγησε την Ισπανία να αλλάξει την ομοθεσία της έτσι ώστε να υπάρχει ένα ελάχιστο όριο επένδυσης σε ε, πολυσχηδή επενδυτικά προϊόντα τα οποία πολλές φορές πρέπει και να απαγορευτούν. Ως προς το ερώτημα υπαριθμών 3, όσον αφορά το μηχανισμό διαιτησίας στα πλαίσια του προγράμματος χρηματοοικονομικής βοήθειας στην Ισπανία για την ε, αναδιάρθρωση των τραπεζών προβλέπεται έτσι ώστε να μην γίνονται παρασωστές ε, πωλήσει, ιδιαίτερα ως προς τα προνομιούχα ομόλογα και μετοχές το 2012. Και με βάση τα δεδομένα των Ισπανικών αρχών φαίνεται ότι μεταξύ 12 και 15 ο μηχανισμός αυτός διαιτησίας έφτασε σε 298.000 αποφάσεις σε σχέση με τους ετούντες, έτσι ώστε να γίνει αποδεκτό το 71% των προσφύγων. Επίσης, ε, το Ταμείο Εγγυήσεων ε, χρειάστηκε να επιστρέψει τα προνομιούχα ομόλογα τα οποία πολίθηκαν ε, κατά τρόπο καταχρηστικό. Ως προς το ερώτημα υπαριθμών 4 σε σχέση με τη νέα ε, νομοθεσία για τα, τις νέες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες θα ήθελα να αναφερθώ την οδηγία για την οδηγία CARP και ΠΡΙΠΣ. Η δανειοδότες θα πρέπει να τονίσουν στους καταναλωτές τους κινδύνους που ενέχονται στα προϊόντα που πολλούν. Και αυτό θα πρέπει να γίνει πριν από την ε, διαδικασία ε, έναρξης εκτέλεσης. Αυτό ορίζεται στην οδηγία ε, για τις υποθήκες, έτσι ώστε να ε, τονίσουν οι πιστωτές του κινδύνους που υπάρχουν. Επίσης, σε σχέση με τα δεδομένα ως προς τις ε, καθυστερούμενες πληρωμές, θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί η σχετική διάταξη σε σχέση με περαιτέρω μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ε, ε, διαδικασίες διακανονισμού. Αυτή τη στιγμή προβάλλονται σε εθνικό επίπεδο οι διαδικασίες ε, διακανονισμού και θα πρέπει τη στιγμή που δεν μπορούν να ανταποκριθούν τα κράτη στα ε, ενυπόθηκα ε, δάνεια θα πρέπει να γίνει μία διευθέτηση με τον δανειοδότη. Η οδηγία διευθέτησης των υποθήκων δεν προβλέπει επαρκώς τη διαδικασία εισαγωγής σε εθνικό επίπεδο. Τώρα, σε σχέση με την λανθασμένη πληροφόρηση ως προς τα προϊόντα, πιστεύω ότι στο μέλλον θα υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση, διότι η οδηγία για την αντιμετώπιση των ε, υποθήκων τονίζει έναν τέτοιο μηχανισμό με βάση και τη συμπεριφορά των ε, επιχειρήσεων και των χρηματοπιστωτικών μέσων έτσι ώστε και οι μεσολαβητές να διεκπαιρεώσουν πολύ σωστά και με διαφάνεια και επαγγελματισμό τις διαδικασίες αυτές έτσι ώστε να μπορέσουν να πληρούν τους όρους αυτούς και άμεση. Αυτό αφορά τις υπηρεσίες επενδύσεων και θα υπάρχει καλύτερη προστασία, επενδυτική προστασία με βάση τα προαπαιτούμενα και τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων έτσι ώστε να μην γίνονται καταχρηστικές πωλήσει. Επίσης υπάρχουν κυβερνητικοί μηχανισμοί έτσι ώστε να μπορέσουν οι επενδυτές να ανταποκριθούν επαρκώς. Η διαδικασία μεταφοράς δεν έχει οριστεί πλήρως, γι' αυτό είναι δύσκολο να πούμε τώρα ποια είναι τα μέτρα τα οποία χρειάζονται περαιτέρω για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής. Ευχαριστώ. Θα αρχίσει η συζήτηση εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων και πρώτη κυρία Σταράς ε, Φεραγούτο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατάρχας ανισχύει πολύ η Ισπανική κυβέρνηση για το ότι έχει γίνει με αυτά τα ε, περίπλοκα προϊόντα ε, με τις προνομιούχες μετοχές, τα ομόλογα που πωλήθηκαν σε πολλούς Ισπανούς και οι εξώσεις που βεβαίως πλήττουν τους πιο ευάλωτους. Στο πρώτο θέμα, πουλήσανε αυτά τα προϊόντα από το 2003 στο 2011 και όταν ήρθε στην κυβέρνηση το Λαϊκό Κόμμα βρήκε την κατάσταση αυτή και πολλές οδηγίες όπως αυτή για τις αγορές το 2008 ε, ή της Βασιλείας το 2011 είχαν ε, προειδοποιήσει την Ισπανική Σοσιαλιστική τότε κυβέρνηση να δράσει, να πάρει μέτρα, να κάνει δράσεις για να ενημερώσει τους πελάτες. Αυτό δεν έγινε. Η Σοσιαλιστική κυβέρνηση τότε ήταν ε, επιπόλαια, μη σοβαρή και στα τέλη του 2011-2012 ε, έγιναν μια σειρά τροποποιήσεις νομοθετικές, όπως πολύ σωστά είπε Επίτροπος, για να μην επανέλθουν ε, σε τέτοια μαζική πώληση αυτά τα προϊόντα στους μικροεπενδυτές και αρχίζει και η διατησία και η διαμεσολάβηση. Πάνω από 71% οι επίτροπος έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Ε, ασχολούμαστε με αυτό το θέμα και το θέμα έχει ε, πλαισιωθεί τώρα για τις εξώσεις. Και πάλι η δική μας λαϊκή κυβέρνηση για πρώτη φορά προστάτευσε τις ευάλωτες ομάδες. Οι πληστηριασμοί και οι εξώσεις του 2014 ήρθαν από στεγαστικά που υπογράφηκαν το 2005 με 2008. Η δική μας λαϊκή κυβέρνηση έφερε μέτρα συγκυριακά για να προστατεύσει του πιο ευάλωτου, όπω πολύ ωραία είπε με αναδιάρθρωση του χρέου, με διαγραφή και ε, με μεταβίβαση αντίπληρωμής. Εμεί το φέραμε αυτό το μέτρο τον Τάτιο του με διαρθρωτικά μέτρα επαναλαμβάνω για να μην επαναληφθούν τέτοια πράγματα στο μέλλον. Και χιλιάδες οικογένειες ε, υποφελήθηκαν. Ακόμα εξακολουθούμε να δουλεύουμε. Ζητάω από τους συναδέλφους να μην κάνουν αυτή τη σημαντική συζήτηση εδώ, προεκλογική συζήτηση. Γιατί δεν αξίζει στα ε, θύματα των ε, εξώσεων αυτή η μεταχείριση. Η πρόεδρο διακόπτη. Λοιπόν, Κυρία Κοζάλες Πένιας, ζητήσατε μπλε κάρτα πριν, αρχίσει, να, πριν ανοίξει το στόμα της η κυρία Σταράς. Έτσι, γαλάζια κάρτα, δεν θέλετε, ναι. Τη δέχεστε. Ναι, έχετε δίκιο, προσπαθήσουμε λίγο να ε, συγκρατήσουμε τη συζήτηση. Κυρία Σταράς, σε, εσείς ζείτε σε μια πραγματικότητα και ο λαός στην Ισπανία σε άλλη. Δεν ξέρω, ίσως γι' αυτό μάλλον ε, το συνδέσατε με τα ε, εκλογικά μέτρα. Υπάρχουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που είπαν ότι η Ισπανική νομοθεσία ε, αντίκειται στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ό,τι αφορά τις εκτελέσεις και τους πληστηριασμούς. Αυτό το λέμε και μια συντριπτική πλειονότητα το 2014 μάλιστα τον Ιούλιο Ισπανή. Θα εξακολουθήσει το Λαϊκό Κόμμα να μας ντροπιάζει εδώ πέρα μέσα χωρίς κανένα λόγο. Ερώτηση είπαμε να κάνετε λέει και είχατε 30 δεύτερα. Madame, c'était une question et vous aviez... Ερώτηση, 30 δεύτερα για ερώτηση. 30 δεύτερα επίση για την απάντηση. Ε, κυρία Σταράση, ευχαριστώ. Μπορεί να σας φαίνεται καλό ή κακό, αλλά τα γεγονότα είναι αυτά που είναι. Από τότε που έμαθε η κυβέρνηση της Ισπανίας ε, την κατάσταση πήρε και διαρθρωτικά μέτρα και συγκυριακά. Ε, και οι ντροπέ και οι πομπέ και τα έσχη είναι δικά σα, δεν είναι δικά μας. Ε, ε, οι σοσιαλιστές και οι δημοκράτες. Τώρα η κυρία Καβεθόν Ρουίς. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Η κρίση κατέδειξε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, μας έδειξε μεγάλα διδάγματα, ότι οι ανυπεράσπιστοι δεν προστατεύονται σωστά ε, απέναντι στις τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στην Ισπανία έχουμε κοινωνική τραγωδία. Είναι γεγονός ότι οι σοσιαλιστές δεν καταφέραμε να δώσουμε απάντηση και δεν το κρύβουμε αυτό. Αλλά δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με αυτή την αδικία που συνεχίζει ε, να βυθίζει σε τραγωδία 107 δισεκατομμύρια ε, δώσανε για τις τράπεζες, για την ε, κεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Ε, Έχουν 171.000 μικροεπενδυτές πληγή και πήραν ε, ένα ε, στα τρία ευρώ, από 30 με 70% ε, συνεχίζουν ακόμα μικροί επενδυτές να είναι παγιδευμένοι. Γι' αυτό η Ισπανική κυβέρνηση τι έκανε. 12 μεταρρυθμίσεις αποσπασματικές και με σαφή διάθεση να δείξουμε ότι όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Δεν έχει καλύψει ούτε κατά διάνοια το πρόβλημα ε, και ε, τι γίνεται με τη μεταβίβαση αντιπληρωμής, τι γίνεται με την κοινωνική στέγη. 3,5 ε, δις είναι σε υποθήκες σε στεγαστικά με καταχρηστικές ρήτρες. Αυτά τα λέει όχι το Σοσιαλιστικό Κόμμα αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το 93-13 η οδηγία αυτή δεν εφαρμόζεται, παραβιάζεται στην Ισπανία σε διάφορα άρθρα. Και από το Μάιο το 2015 υπάρχει η απόφαση που ορίζει ρητά ότι ε, τα όσα κάνει η Ισπανική κυβέρνηση είναι τελείως ανεπαρκή. Γι' αυτό δεν θέλουμε εμβαλωματικές δράσεις, ε, χρειαζόμαστε μια γενική ε, απάντηση για να μην εμπέζουμε το λαό. Παρακαλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια σοβαρή ανάλυση για το πόσο ε, τηρείται ο νόμος ή όχι και ποιες είναι οι καταρχικές ρήκτες και να προστατεύονται οι μικροί επενδυτές που εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Πολλά πράγματα έχετε να πείτε βλέπω σε αυτό το θέμα, αλλά σας παρακαλώ να τηρείτε το χρόνο σας. Ιδίω όταν μιλάτε εκ μέρου των ομάδων. Τώρα το λόγο έχει το ΙΣΙΕΡ ο κύριο Μαριά. Για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, η νομοθεσία για τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφοροποίηση στου όρου για την προστασία του καταναλωτή και στο διακανονισμό του χρέου στην ισπανία αλλά και στην ελλάδα πολλές φορές δεν υπήρξε η κατάλληλη ενημέρωση των δανειοληπτών από τις τράπεζες και οι όροι των συμβολέων παραβιάζουν τα δικαιώματα των δανειοληπτών ως καταναλωτών. μετά την χρηματοοικονομική κρίση επιδεινώθηκε η κατάσταση στην ισπανία με αποτέλεσμα τουλάχιστον 700.000 πολίτες να είναι θύματα των δανείων υψηλού κινδύνου ενώ τα τελευταία έξι χρόνια έχουν καταγραφεί πάνω από 350.000 εξώσεις. ταυτόχρονα οι κατοικίες που βγήκαν στο σφυρί επανήλθαν στην ιδιοκτησία των τραπεζών οι οποίες ως γνωστόν έχουν διασωθεί από τα χρήματα των ίδιων των πολιτών της ευρωπαϊκής ένωσης. στην ελλάδα τα κόκκινα στεγαστικά δάνεια έφτασαν τα 21 δισεκατομμύρια ευρώ εκεί οι τράπεζες άρχισαν να πολλούν τα κόκκινα δάνεια στα γνωστά κοράκια τη παγκόσμια αγορά, στα επιθετικά hedge funds που ετοιμάζονται να βγάλουν στο σφυρί αντί πινακίου φακής στα σπίτια του ελληνικού λαού. μάλιστα με το μνημόνιο τρία διαμορφώνονται και διαδικασίες εκπρές για τους πληστηριασμούς. πάνω από 500.000 έλληνες δανειολήπτες κινδυνεύουν πλέον να χάσουν τα σπίτια τους. επίσης 70.000 έλληνες που έχουν συνάψει ενυπόθηκα δάνεια σε ελβετικό φράγκο κινδυνεύουν και αυτοί να χάσουν τα δικά τους σπίτια για τον λόγο αυτό ως μέλος της επιτροπής αναφορών ζητώ η ευρωπαϊκή επιτροπή σε συνεργασία με την κεντρική τράπεζα να πάρουν μέτρα για την προστασία της πρώτης κατοικίας και να σταματήσουν οι πληστηριασμοί των σπιτιών στην ελλάδα και την ισπανία. ευχαριστώ. κυρία κυρία Ευχαριστώ για τις λεπτομερείς εξηγήσει που μας δώσετε σήμερα. Μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για το ότι μία προφορική ερώτηση με ψήφισμα φτάνει στην Ολομέλεια. Είναι μεγάλο νέο, γιατί δεν ήθιστε η Επιτροπή Αναφορών, η οποία είναι ουσιαστικά το παράθυρο των πολιτών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δράμα αυτόν τον τρόπο. Και νομίζω ότι από το 2012 και μετά από τις δικτυμαρικές δεν είχαμε τέτοια δυνατότητα. Είμαστε εδώ σήμερα λοιπόν γιατί πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες θύματα καταχρηστικών ρητρών και πρακτικών θύματα των προνομιούχων μετοχών. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς είναι, μπορεί να είναι εκατομμύρια, ή δεκατομμύρια. Πάντως στην Επιτροπή Αναφορών πρέπει να ξέρετε ότι δεκάδες τέτοιες αναφορές παίρνουμε συνέχεια από Ευρωπαίους πολίτες που βλέπουν ότι έχουν πληγεί τα θεμελιώδη τους δικαιώματα στην Ισπανία. Πρόκειται λοιπόν για μια ευρωπαϊκή υπόθεση. Είναι Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν στην Ισπανία και τους οποίους πρέπει να προστατεύσουμε. Και η, και η Επιτροπή Αναφορών πρέπει να κρατάει ανοιχτέ τι αναφορέ του και να φροντίσει να υπάρξει μια συμφωνία. Γι' αυτό και βρισκόμαστε εδώ. Οι Ισπανοί καταναλωτέ είναι σε μια κατάσταση όπου βρίσκονται προστάτευτοι, ακάλυπτοι. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το είπε αυτό. Και αυτό ακριβώ και αιτιολογεί και την παρέμβαση των Ευρωπαϊκών Αρχών. Και μιλάμε και για ένα ευρωπαϊκό ζήτημα, γιατί πρόκειται για κακή εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών. Στην πραγματικότητα, οι αναφορές αυτές καταγγέλουν την ε, κακή ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο οδηγιών για τα ανυπόθηκα δάνεια ή για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που πρόκειται για επενδυτικά προϊόντα και για προνομιούχες μετοχές μέσω καταχρηστικών ρητρών και πρακτικών σε βάρος των καταναλωτών Πιστεύω ότι παρόλο που ακόμα υπάρχουν αδυναμίες στην μεταφορά των ευρωπαϊκών ε, οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, η προσπάθεια γίνεται και υπάρχει βελτίωση. Δεν έχει σημασία σε ποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνονται όλα αυτά. Σημασία έχει να καταγγέλουμε όταν κάτι πάει στραβά και να φροντίζουμε να διορθώνουμε τα πράγματα για να προστατεύουμε τους πολίτες και να τους διαφαλίζουμε τη ρίση των δημιουργών τους δικαιωμάτων. Αυτά και στη γραμμή των όσων είπε η κυρία Γιούροβα. Δηλαδή πρέπει να εποπτεύουμε και να φροντίζουμε να μην ξανασυμβεί ποτέ το ίδιο. Ευχαριστούμε. Η κυρία Βαλίνα τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Από την αρχή της ε, κρίσης στην Ισπανία 590.000 εξώσεις έλαβαν χώρα και Πρόκειται βέβαια για πάρα πολλά θύματα των προνομούχων μεταχών. Οι ίδιοι χάνουν τα χρήματά τους από τις τράπεζες συγχρόνως εξαιτίας της κρίσης. Σημειώνεται οι μισθοί τους, είχαν λιγότερες δυνατότητες εκπαίδευσης κτλ. Και επιπλέον ε, έχουμε χιλιάδες κενές κατοικίες. Πάρα πολλές περιπτώσεις επίσης διαφθοράς εντοπίστηκαν που καταστρέφουν τις ε, το τραπεζικό τομέα. Γι' αυτό λοιπόν και σήμερα εμείς μεταφέρουμε τις φωνές χιλιάδες ανθρώπων για δικαιοσύνη, για τα θεμελιώδη τους δικαιώματα. Δικαιώματα όπως είναι το δικαίωμα στην κατοικία. Δικαιώματα προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχει μια νομοθεσία κατά των χρηματοπιστωτικών αυτών απατών. Ευχαριστούμε για δύο λεπτά ο κύριος Τερικάμπρας εκ μέρους των Πρασίνων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή Αναφορών, στην οποία ανήκω, απαντώντας ε, στις αιτήσει των πολιτών, μίλησε για τη λανθασμένη εφαρμογή ε, από τη χώρα μου του κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό οδήγησε σε ένα μεγάλο κοινωνικό δράμα. Σύμφωνα με τα δεδομένα, μεταξύ 8 και 12 στην Ισπανία είχαμε 170.000 εξώσεις και μεταξύ 12 και 14 είχαμε 100.000 ε, εκτελέσεις της απόφασης ε, πληστηριασμού. Ε, άρα είναι σαφές ότι υπάρχουν καταχρηστικές ρήτρες και δεν μπορούμε να διασώζουμε τράπεζες τη στιγμή που δεν θα βοηθήσουμε τις τους καταναλωτές. Ένα 32% ε, στη χώρα των Βάσκων... Ε, ε, στις κάτω χώρες ένα 32% χορηγείται για την κατοικία, ενώ στη δική μου χώρα ένα 1 με 2%. Άρα θεωρώ ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε πολυσχηδή χρηματοπιστωτικά μέσα. Γι' αυτό θα ήθελα, κυρία Επίτροπε, καταρχήν ε, να ζητήσουν τα ρυθμιστικά όργανα να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη συγκεκριμένα ρυθμιστικά πλαίσια λειτουργίας. Επίσης, ο καταναλωτής να μπορεί να παραδώσει την κατοικία ως μέρος της αποπληρωμής μέσα στα πλαίσια της απόδοσης ή αποπληρωμής του χρέους επίσης να αντικατασταθεί η οδηγία που ισχύει εδώ και 22 χρόνια ε, με μια πραγματικά να προστατεύει τους καταναλωτές. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό. Η κυρία Εύη. Ευχαριστώ. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια ισπανική υπόθεση, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση σήμερα για να προσδώσουμε σημασία σε δεκάδες αιτήσει που αναφέρονται σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και απαράδεκτο που αφορά ε, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους μέσα στα πλαίσια αυτών των αναφορών που λάβαμε. Πρόκειται για ένα θέμα που δεν αφορά μόνο την Ισπανία και αναφέρομαι στην υπερεξουσία των ε, τραπεζών που διαθέτουν προϊόντα υψηλού κινδύνου σε καταναλωτές. Αυτό είναι απαράδεκτο, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε το συντομότερο δυνατόν να προστατευτούν οι καταναλωτές και αυτό αφορά μια γενικότερη πολιτική υπεράσπισης των καταναλωτών. Άρα στο ψήφισμά μας θα πρέπει να τονιστεί το δικαίωμα στην πρώτη κατοικία και να το λάβει υπόψη η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνονται οι τοποθετήσει των πολιτικών ομάδων με μονομένη τώρα. κύριο Μάτο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Όλοι γνωρίζουν ότι αυτή η συζήτηση δεν θα έπρεπε να γίνεται εδώ αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο επειδή βασικά και ουσιαστικά είναι εθνικό θέμα, όπω επανειλημμένα ακούστηκε, αλλά επειδή ε, φάνηκε κιόλα μετά από τι τοποθετήσει που ακούσαμε. Και το γνωρίζουν πολύ καλά κάποιες Ισπανίδες ε, αριστερές συνάδελφοι εδώ παρούσες. Δημόσια χρησιμοποιούν αυτό για ίδιους σκοπούς και μάλιστα εκλογικούς. Και δεν το λέω εγώ, το λένε εκείνες και γραπτός μάλιστα. Έχετε δίκιο, η αριστερά ε, κάνει μία χρήση ε, τελείως αποκρουστική και απορριπταία των δεινών που πλήττουν τους πολίτες. Η κυβέρνησή μας ανησυχεί γι' αυτό και ανησυχούσε και θα έπρεπε να είχε λυθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση η οποία το αγνόησε. Το αντίθετο πήραν νομοθετικά μέτρα τώρα και ε, έχουν κάνει μια διατησία υπέρ των πληγέντων. Αυτό το αναγνωρίζει και η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά αυτό εσά δεν σας ενδιαφέρει, πολλές από εσάς. Σας ενδιαφέρει ποιος θα βγάλει το πρώτο δελτίο τύπου, ποιος θα κάνει τον περισσότερο θόρυβο και τη φασαρία και πώς θα το αξιοποιήσετε αυτό. Η Ισπανική κυβέρνηση εντατικά εργάζεται για να λυθεί το πρόβλημα εκείνων που έχουν δυσκολία να πληρώνουν τις δόσεις τους. Ε, χιλιάδες οικογένειες στην Ισπανία. Είναι πολύ οδυνηρή η κατάσταση, χωρίς καμιά αφιβολία, αλλά αυτό ανάγεται έτη πριν το 2008. Η δική μας κυβέρνηση με θάρρο και αποφασιστικότητα ελαστικότητα το αντιμετώπισε με νομοθετικά μέτρα, με βοήθεια προς τους πληγέντες που αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Πάνω από 30.000 οικογένειε ήδη έχουν επωφεληθεί από τα διαρθρωτικά και τα συγκυριακά μέτρα που πήραμε. Το Λαϊκό Κόμμα. Αλλά μην ξεχνάτε, αυτοί που σήμερα υποφέρουν αξίζουν πολύ περισσότερα από ένα τίτλο στι Εφημερίδε. Ευχαριστώ πολύ. Δέχεστε μπλε κάρτα κύριε Μάτο. Από την κυρία Τόρες Μαρτίνες. Μάλιστα, δέχομαι. 30 δεύτερα. Επονίδιστο είναι, τι, έσχος, δεν, τι, αχαρακτήριστο. Τι είναι αυτά που λέει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ε, πραγματικά μας έχει γεμίσει αγανάκτηση και αποτραπιασμό. Δεν τρέπεστε με την αδράνειά σας, με την παθητικότητά σας απέναντι στις άλλες ομάδες και στους Ισπανούς, με τις εξώσεις πέρα από τα προεκλογικά δύο μήνες σας μένουν, δύο μήνες για να επανακτήσουμε ε, τα δικαιώματα των ανθρώπων, για να σας διώξουμε από τους θεσμούς που μας έχετε καταλυστεύσει και καταντροπιάσει. Ευχαριστώ κύριο Μάτο. Ήδη ε, απαντάει. Ζήτησε γαλάζια κάρτα πριν ανοίξω το στόμα μου. Οπότε καταλαβαίνετε τι με περίμενε. Τι, τι ήθελε, δημαγωγία, λαϊκισμό και ακτιβισμό. Αφήστε σε δύο μήνες οι πολίτες να αποφασίσουν ε, και θα πάει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Curtin Darling, in minute. Για ένα λεπτό, κυρία Curtin Darling. Ευχαριστώ. Στην Επιτροπή Αναφορών είμαι και εγώ μέλος και επικεντρωνόμαστε στον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τους πολίτες στην Ισπανία τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά και σε άλλες χώρες όταν πλήττονται θεμελιώδη δικαιώματά τους. Βρετανοί ζουν στην Ισπανία και πολλοί από αυτούς έχουν ανυπόθηκα δάνεια. Για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των ε, πολιτών λοιπόν και για να μπορούν να συνεχίσουν να παίρνουν ανυπόθηκα δάνεια θα πρέπει όλες οι χώρες να πιέσουν τις τράπεζες να δίνουν κατανοητές και ορθές πληροφορίες στους καταναλωτές. Η οδηγία για τα ανυπόθηκα δάνεια θα βοηθήσει να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια στην εσωτερική αγορά και θα πρέπει όμως να προσφέρει και μεγαλύτερη προστασία για τους καταναλωτές. Οι ευρωπαϊκοί πολίτες κάνουν έκκληση για δράση μέσω των αναφορών αυτών που μας στάνουν. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πρέπει να ακούσουμε την έκκλησή τους και να φροντίσουμε να προστατεύονται τα δικαιώματά τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για δυόμιση λεπτά η κυρία Μπιλμπάου Παραντικά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ την Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών και τα μέλη της Επιτροπής αυτής για τις προσπάθειες που κάνουν προκειμένου τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να προσφέρουν ελπίδα και λύσεις σε πολλές οικογένειες. Η, το υπερβολικό θράσος, κάποιες εμπορικές πρακτικές, καταχρηστικές και μια άδικη νομοθεσία και ανεπαρκής και ένα ε, μοντέλο ανάπτυξης κερδοσκοπικό οδήγησε στα δράματα αυτά που αντιμετωπίζουν τόσοι πολίτες με εξώσεις κλπ. Δεκάδες χιλιάδες οικογένειες έχουν χάσει τη, τα σπίτια τους, τη δουλειά τους. Άλλοι τόσοι έχουν προσωπικά δράματα. Αγόρασαν, ε, πήραν ενυπόθηκα δάνεια για τα παιδιά τους και οδηγήθηκαν σε καταστάσεις πραγματικά κατεπίγουσες κοινωνικά και ανθρωπιστικά. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Επίτροπη Βρυξέλλες πρέπει να υποχρεώσουν τις πανικές αρχές τις, ε, την ιδεοντολογία των τραπεζών να την ε, καταστήσουν υποχρεωτική. Διότι πρέπει να έχουν ισότητα εκείνοι οι οποίοι παίρνουν δάνεια και εκείνοι οι οποίοι τα δίνουν. Σε περίπτωση μάλιστα δυναμίας εξόφλησης αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τα διάφορα δράματα έχουν να κάνουν με το ότι οι καλοί τυπίστοι καταναλωτές πήραν τα δάνεια που τους πούλησαν αδίστακτοι. Ούτε όλε οι οικονομίες, ούτε όλα τα οικονομικά ιδρύματα δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο. Το πρώτο τρίμηνο του 2013, 0,20% των υποθηκών για κατοικίε ανάμεσα στο 2003 και το 2014 προχώρησαν και έφτασαν στα δικαστήρια στην Ισπανία. 17.786 πιο συγκεκριμένα. Η χώρα των Βάσκων με 0,02% είναι η περιφέρεια της Ισπανίας, με απόσταση από τις υπόλοιπες, που έχει πάρα πολύ χαμηλό δίκτυ τέτοιων δικαστικών υποθέσεων. Οι πρακτικές διαπραγμάτευσης βοήθησαν και μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς προκειμένου να μειωθούν οι τραγωδίες αυτές που αντιμετωπίζουν τόσοι άνθρωποι οι οποίοι υφίστανται εξώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Κούνεβα, παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εκατοντάδε χιλιάδε πολίτε στην Ισπανία, την Ελλάδα και άλλα κράτη-μέλη όπω τη Βουλγαρία εξαπατήθηκαν στην προσπάθεια του να αποκτήσουν δικαίωμα στην κατοικία με τραπεζικό δάνειο. Δικαίωμα αναγνωρισμένο ω αναφέρετο ήδη από το 1948 στην ιδρυτική διακήρυξη του ΟΗΕ. Και όμω, 67 χρόνια μετά, η Κομισιόν κάνει πω δεν ακούει. Και α έχουμε σημαντικά θεσμικά εργαλεία ελέγχου, όπω οι οδηγία προστασία των καταναλωτών και η απόφαση του Ευρωδικαστηρίου για την υπόθεση Αζή. Οι 398.000 εξώσει από το 2008 στην Ισπανία δείχνουν ότι οι νόμοι που προστατεύουν τους δανειολήπτες από την κατάχρηση των τραπεζών δεν ελέγχονται και οι καταγγελίες που μας έρχονται από τη Βουλγαρία μας προβληματίζουν εάν η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή υποπτεύει σωστά. Στην Ελλάδα τα κόκκινα δάνεια μοιάζουν με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί. 260.000 δανειολήπτες στο κόκκινο, οι περισσότεροι άνεργοι χωρίς εισόδημα, αγωνιούν για το εάν τα έχουν τη τύχη των Ισπανών μετά την λήξη του capital control, ίσως και νωρίτερο όταν οι πρόσφυγες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στο έλεος του πολέμου και αναζητούν σωτηρία στην καρδιά της Ευρώπης η ίδια δεν μπορεί να εξασφαλίσει την κατοικία των πολιτών της. Ας δείξει λοιπόν η Κομισιόν ότι δεν τους βλέπει σαν ψηλά γράμματα των τραπεζικών συμβάσεων, να ασκήσει σοβαρά έλεγχο και να δώσει ανάσα ζωής στα τίματα του τραπεζικού κατεστημένου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σουρτάσουν για ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε του ΕΛΚ, ήδη είστε καταδικασμένοι πολιτικά με αυτό το δράμα, το ανθρώπινο. Και ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες υπογραφές έχουν μαζέψει πολίτες και τους ε, αγνοείτε. Σας λέει η Επίτροπος ότι ο Ισπανικός νόμος ε, ε, δεν ε, σέβεται την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτά τα πράγματα δεν μπορείτε να τα λέτε. Κυρία Επίτροπε, θέλω να σας πω το εξής. Υπάρχουν ενδείξεις ότι και στο αστικό δίκαιο και στα θέματα που αφορούν τις υποθήκες δεν γίνεται σεβαστή η ευρωπαϊκή νομοθεσία παρά τις αλλαγές στην νομοθεσία και το 2013 και το 2015. Τι να περιμένουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ε, έρχονται ε, στην Επιτροπή Αναφορών και μας λένε ότι έχουν διαρθρωμένο διάλογο η Κομισιόν με την κυβέρνηση. Και τι κάνουμε στο μεταξύ με τους, 68.000 που τους έχουν κάνει πληστηριασμό. Θα περιμένουν το 2016 και άλλες χιλιάδες φέτος. Είναι ανθρώπινα δράματα. Κάντε κάτι. Εάν δεν υπάρχει αντιμετώπιση από την Ισπανική νομοθεσία νομοθεσία. Κάντε κάτι εσείς, αναλάβετε δράση. Παρακαλώ, κυρία Γκίλ. Η μεγάλη κρίση ενυπόθηκων δανείων στις ΕΠΑ το 2008 ε, μετακυλίστηκε στην Ευρώπη γιατί ε, ακριβώς ε, έγιναν δανειοδοτήσεις που ήταν εντελώς ανεύθυνες και αυτό το είδαμε και στην Ισπανία διότι ε, πολύ ε, δυστυχώς και στην Ισπανία δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν και δέχομαι την κατάστασή τους. Θα πρέπει να μην γίνουν εξώσεις, ιδιαίτερα αυτών που έχουν ανάγκη, δηλαδή τους υπερήλικες και τους νέους με οικογένεια. Το 2011 η Κομισιόν ε, δημιούργησε μία νέα οδηγία για την αντιμετώπιση της ενυπόθηκης αγοράς με ε, προστασία έναντι κινδύνου. Αυτό όμως θα πρέπει να εφαρμοστεί προς όλα τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ε, μία πολύ σωστή δανειοδοτική πολιτική χωρίς κινδύνους. Για δυόμιση λεπτά η κυρία Πακαζόρντου Ρουίθ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Και ευχαριστώ κυρίως την Πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών, γιατί με τις προσπάθειές της αντιμετωπίζονται οι αναφορές τόσων πολιτών. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν και για τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε. Οι πολίτες είμαστε και καταναλωτές και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη σε εκείνους που μας παρέχουν υπηρεσίες που είναι βασικές για τη ζωή μας. Και οι τράπεζες αποτελούν μέρος της κατηγορίας αυτής. Για να είμαστε ξεκάθαροι, σε αυτήν την ολομέλεια αρχίζουμε να εξετάζουμε διάφορα θέματα που απασχολούν τον κόσμο και στην Ισπανία, αλλά και όχι μόνο δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίους πολίτες. Για παράδειγμα, το πιο τραγικό είναι η περίπτωση αυτών των περίπλοκων χρηματοπιστωτικών προϊόντων που είχαν σαν ε, αποτέλεσμα να πληγούν εκατοντάδες χιλιάδες ε, πολίτες. Θέλουμε απαντήσεις και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να μας τις δώσει σύντομα. Και στηρίζουμε οποιαδήποτε τρόπο οπουδήποτε πρωτοβουλία η οποία θα βοηθήσει να σταματήσουν αυτές οι καταχρηστικές πρακτικές και οτιδήποτε άλλο κάνει καταστά τους καταναλωτές απροστάτευτους και δύναμους. Στηρίζουμε έναν ακέραιο οικονομικό τομέα. Υποστηρίζουμε υπεύθυνε πολιτικές χωρίς διαφθορά. Η απάτη με τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα φάνηκε γιατί εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες κατάλαβαν έτσι τους το εξήγησαν ότι επρόκειται για σταθερής απόδοσης προϊόντα, ενώ τελικά επρόκειτο για κειμενόμενης απόδοσης προϊόντα. Αυτή ήταν η απάτη. Για μένα προσωπικά, εμένα μου ζήτησε ένας ε, χείρος βοήθεια. Η γυναίκα του είχε δολοφονηθεί σε μια τρομοκρατική επίθεση και είχε αγοράσει προνομιούχες μετοχές με την αποζημίωση που είχε πάρει για τη δολοφονία της γυναίκας του χωρίς να έχει καταλάβει τι έκανε τελικά. Έπειτα υπάρχουν οι τέσσερις οδηγίες που δεν εφαρμόζονται σωστά. Όμως, από την άλλη μεριά, χρησιμοποιήθηκε και έγινε πολιτική εκμετάλλευση αυτή τη υπόθεση με τα μυευτήρια. Το κόμμα μας τον Απρίλιο του 2013 πήγε στα δικαστήρια για να αποδοθούν ευθύνε. Ευχαριστούμε. Αλβιόλ Μπουδμαν τώρα. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι κάνουμε λάθος ε, γιατί η ουσία αφορά την ε, Σαταντέρ και και την και εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για ληστρικούς οργανισμούς που κατακλέβουν τον κόσμο. Δηλαδή μιλάμε για τραπεζικούς οργανισμούς οι οποίοι, οι οποίοι στην ουσία υπηρέτησαν την πολιτική εξουσία ε, γιατί οι κυβερνήσεις Θαπατέρο και Ραχώη στην ουσία δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να υποστηρίξουν όσους έκαναν εξώσεις και απάτες. Μιλάμε για 71 δις ευρώ άμεσες ενισχύσεις για την υποστήριξη των τραπεζών. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μιλήσω για την μεγάλη... Νομίζω ότι έχει σημασία να υποστηρίξουμε τη μεγάλη αυτή πλατφόρμα η οποία υποστήριξε ε, εκείνους οι οποίοι βρέθηκαν σε κατάσταση έξωσης. Μαραγάλ, κατανοώ σήμερα την θέση του Λαϊκού Κόμματος. Και καταλαβαίνω ότι αυτό το ζήτημα έφτασε στην Ολομέλεια μετά από πολλούς πολίτες και αρχές οι οποίες δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε μια πραγματικότητα που τους αφορούσε όλους. Δηλαδή μια Ευρώπη η οποία δεν μπορεί να ε, καταπολεμήσει την αδικία Δυστυχώς ε, ε, χρειάστηκε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο και οι κυβερνήσεις μας, τα χρηματοπιστωτικά ε, όργανα δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν, γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Μιλάμε για τα ενυπόθηκα δάνεια για την κατοικία και μιλάμε και για τα ε, προνομιούχα ομόλογα τα οποία έχουν δελεαστικό χαρακτήρα αλλά τα οποία προωθούνται ατιμωρητοί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαυρίδης παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μια αξιόλογη δράση της Επιτροπής Αναφορών. Εάν αντικαθιστούσαμε όμως τη λέξη Ισπανία με τη λέξη Κύπρο, όλα τα υπόλοιπα ισχύουν και κατά πολύ χειρότερα και η αναποτελεσματική εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και η αδράνεια που παρατηρείται μπορεί η απόλυτη αριθμή στην περίπτωση της κύπρου να είναι μικρή αλλά ως ποσοστό σε άλλο κράτος μέλος μεγάλο θα ήταν τεράστια. και αυτό αφορά και τα έγγραφα ειδικά προς τους δανειζόμενους όπου υπάρχουν στην κύπρο μέχρι σήμερα και χρησιμοποιούνται συστηματικά και μαζικά καταχρηστικές πρόνοιες και καταχρηστικές πρόνοιε τέτοιε μάλιστα που είτε είναι στον κατάλογο τη Ευρωπαϊκή Οδηγία, είτε έχουν αξιολογηθεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο ω τέτοιε παράνομε. Επίση, άλλο τεράστιο πρόβλημα είναι τα λεγόμενα αξιόγραφα τα οποία πουλήθηκαν σε ανυποψία του, παραβιάζοντα την ευρωπαϊκή νομοθεσία ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας οδηγήθηκε στον μαρασμό και στην κοινωνική αποξένωση και στην αυτοκτονία ακόμη. γι' αυτό λοιπόν δεν μιλάμε μόνο για συμφωνίες. και μια εισήγηση προς την επίτροπο εξώδικος μηχανισμός επίλυσης τραπεζικών διαφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο νομίζω θα βοηθήσει το πρόβλημα. Ευχαριστώ, Ο κύριος Σεμπαστιά, επίσης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Μπορεί να ενοχλεί αυτό ορισμένου, αλλά είναι απολύτω ευρωπαϊκό. Είναι καταχρηστικές πρόνοιες των ε, τραπεζών της Ισπανίας που καλύπτονται ε, και καλυπτόντουσαν. Ε, μισό εκατομμύριο οικογένειες είναι Ευρωπαίοι που έχουν καταδικαστεί στην Ένδια. Γιατί το σκάνδαλο αφορά πολίτες για τα προνομιούχα επίση και τα ταμεία διάσωση 107 δισεκατομμύρια πήραμε για να σώσουμε τις ίδιε τράπεζες και αυτά ευρωπαϊκά κονδύλια είναι και με αυτά σώσαμε τις τράπεζες και ε, ε, βάλαμε αυτές τις τρομερές πολιτικές λιτότητας που πλήττουν τόσο σφοδρά τον κόσμο. Υπάρχει και αποφάση δικαστηρίου που δείχνει ότι είναι ε, παράνομη η δράση της ισπανικής κυβέρνησης και αυτή η ευρωπαϊκή απόφαση είναι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θα πρέπει η Ευρώπη, κυρία Επίτροπε, να δράσει, να σταματήσει αυτό το υποτίθεται νομικό καλοπισμό που κάνει η ισπανική κυβέρνηση δράση. η Ευρώπη δεν αξίζει να έχει αυτό το ρόλο που όλοι εμείς εδώ θέλουμε να της αποδώσουμε. Ευχαριστώ κύριο Φρουντσούλ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό αριθμό αναφορών που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ε, καταχρηστικές ε, ρήτρες που ε, διακατέχουν τα υπόθηκα δάνεια, που διέπουν τα υπόθηκα δάνεια και αυτό θα πρέπει να τεθεί ε, ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως ε, τέθηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου με βάση τη διαδικασία επί παραβάση. Είναι πολύ κρίσιμη η κατάσταση στην Ισπανία. Από το 2008, 700.000 Ισπανοί πολίτες έπεσαν θύματα οικονομικής απάτης και 400.000 βγήκαν από τα σπίτια τους. Νομίζω ότι οι Ισπανικές αρχές θα πρέπει να λάβουν όλα τα μέτρα για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Ε, Φερνάντες, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την Πρόεδρο και τη συνάδελφο Σολετάδ Καμπεθών που εργάστηκε πολύ σκληρά τις τελευταίες εβδομάδες για να υποβάλει αυτή την ερώτηση προς την Κομισιόν. Τα σκάνδαλα τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας ήταν πολλά. Μιλάμε για τα ενυπόθηκα δάνεια, όπου δεν υπήρχε δυνατότητα διαπραγμάτευσης μεταξύ καταναλωτών και τραπεζών και μιλάμε και για τα προνομιούχα ομόλογα, τα οποία έπληξαν πολλούς νέους και γέρους στην χώρα μου. Και Τις τελευταίες εβδομάδες συζητήθηκε το θέμα και γι αυτό, ευρέως και γι' αυτό θα πρέπει η Επιτροπή να δημιουργήσει έναν νόμο δεύτερης ευκαιρίας έτσι ώστε να μπορέσουν οι ε, δανειολήπτες να αντιμετωπίσουν ε, την επώδυνη κατάστασή τους σε μια χώρα που η κυβέρνηση δεν δράει επί της ουσίας. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Πόλτσεκ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ σε αυτά που υπόθηκαν πέρα από την εθνική συζήτηση. Μερικές φορές η αλήθεια είναι ότι η συζήτηση έγινε σε καθαρά εθνικό επίπεδο. Πάντως η έλλειψη διαφάνειας μάλλον η διαφάνεια, οι εγγυήσει, η προστασία των καταναλωτών, αυτά είναι πράγματα τα οποία αξίζει να αναφέρονται σε αυτή τη συζήτηση και είναι βέβαια αλληλένδετα με το θέμα που εξετάζουμε εδώ. Αυτά που είπαμε για τα, τις οικονομικές πληροφορίες, την ενημέρωση που πρέπει να έχει ο καταναλωτής που παίρνει ένα υπόθεκο δάνειο, αυτό είναι πολύ σημαντικό ο αναλφαβητισμός σε τέτοια ζητήματα είναι ζωτική σημασία. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να μπορεί να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά όχι να αναμειγνύεται στα εθνικά ζητήματα. Ευχαριστώ, κύριε Ζάου και Τέντο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ήμουνα πέντε χρόνια στην Ισπανική κυβέρνηση και δεν με ενδιαφέρει να αναγνωρίσω το ότι η Ισπανική νομοθεσία δεν ε, προσαρμόζεται. Δεν με ενδιαφέρει η αναγνώριση το ότι τα χρηματοπιστωτικά μας προϊόντα δεν ήταν καλά, τα δικά μας ή άλλων. Να το αναγνωρίσω. Βεβαίως. Αυτό όμως το οποίο είναι ζωτική σημασίας είναι ότι λέμε ότι η κυβέρνησή μας τέσσερα χρόνια αργότερα τι λέτε, λέτε ότι οι προηγούμενοι φταίγανε, ενώ είσαστε τέσσερα χρόνια στην κυβέρνηση. Αυτό είναι που ενοχλεί. Αλλιώ, εντάξει, να τα αναγνωρίζουμε τα πράγματα. Να πούμε ότι ήταν κακή νομοθεσία, ότι είχε κενά, ότι είχε καταχρηστικέ ρήτρε που δεν θα έπρεπε να υπήρχαν. Και αυτό θέλω να κάνει η Επιτροπή. Αλλά το Λαϊκό Κόμμα δεν μπορεί να λέει ότι εκείνοι τα έκαναν όλα καλά και για όλα φταίγανε οι προηγούμενοι. Ευχαριστούμε. Γιακοβίτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι εμείς ε, λέμε ε, ε, ότι θέλουμε να ρυθμίζουμε τα πάντα. Ποιες γραμματοσυρές θα χρησιμοποιούμε, τι θα γράφουν οι κονσέρβες, τι θα γράφουν οι ετικέτες. Ενώ όταν πρόκειται για χρηματοπιστωτικά προϊόντα δεν ρυθμίζουμε την κατάσταση στην Ισπανία, Ελλάδα, Κύπρο αλλά και στην Κροατία. Ε, τα στεγαστικά ε, δάνεια έχουν καταστρέψει κόσμο. Ήταν κλασική περίπτωση ε, τραπεζικής απάτης. Τα πάντα, ξέρετε, είναι τα ψηλά γράμματα των συμβολέων και δεν υπάρχουν ρυθμίσεις για ποια, το ποια γραμματοσυρά θα χρησιμοποιείται εκεί στις συμβάσεις και στα συμβόλαια που υπογράφουμε όταν παίρνουμε δάνεια. Ενώ επαναλαμβάνω, για τις ετικέτες στις κονσέρβες έχουμε ρυθμίσει και το μέγεθος της γραμματοσυράς. Θα πρέπει να τερματιστεί αυτή η καταχρηστική ε, πρακτική και η απάτη. Ευχαριστώ. Η κυρία Σέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε η καταπολέμηση των εξώσεων και ε, η προστασία των πληγέντων δείχνει ποια είναι η τραγωδία χιλιάδων οικογενειών που χάσανε ή κοντεύουν να χάσουν τα σπίτια τους. Εξακολουθεί αυτό. Τους έχουν κλέψει η τράπεζα οικονομίες μια ζωή ολόκληρη ή τη ζωή τους την ίδια. Αυτό έγινε με συνενοχή και ε, ανοχή της ισπανικής κυβέρνησης. Είδαμε πώς προστάτευσαν τις τράπεζες και ε, ποινικοποιούν, καταστέλουν και ε, τρομάζουν τον κόσμο που θέλει να δικαιωθεί. Είδαμε εξώσεις, βίες οικογενειών από τις ε, από τα σπίτια τους και πώς τους διώκει η αστυνομία. Τώρα έχει έρθει η ώρα να δικαιωθούν. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τερματίσουν τις καταχρήσεις των τραπεζών ε, και να σταματήσει η πολιτική λιτότητα. Η Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Γιούροβα. Παρακαλώ, εξ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Όπως είπα και πριν, η κοινοτική νομοθεσία θα πρέπει να μεταφερθεί και να επιβληθεί στα κράτη-μέλη έτσι ώστε ο νόμος να ανταποκριθεί στο στόχο του. Επίσης θα πρέπει να δίνονται περισσότερες και σωστότερες ε, πληροφορίες στους καταναλωτές. Συμφωνώ ότι τα προληπτικά μέτρα είναι ακόμα πιο σημαντικά και πιο ε, αποδοτικά από τον σκληρό νόμο. Αλλά είναι κάτι που επιβάλλεται. Όπως σας είπα, αναλύουμε τις απαντήσεις των Ισπανικών αρχών που λάβαμε τον Ιούνιο, ε, ιδιαίτερα σε σχέση με τον νόμο που διέπει τα ενυπόθηκα δάνεια δάνεια. Επίσης, ε, αν η απάντηση δεν είναι ικανοποιητική, τότε θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα αμελητή. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι θα υπάρξει προστασία των καταναλωτών. Όταν οι καταναλωτές άγονται ενώπιον του δικαστηρίου θα πρέπει να την χάνουν προστασίας όπως ορίζει και η πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και Πολλοί από εσά ε, ε, μιλήσατε για την ε, ενδεχόμενη αφαιρεγγιότητα και πώς διέπει το όλο πλαίσιο λειτουργίας και αντιμετώπιση των ενυπόθηκων δανείων. Θα ορίσουμε τον κανονισμό περί αφαιρεγγιότητας του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ. Λίγη η συζήτηση.